θέμα της μέσης διάταξης για απόψε η έκθεση ΣΑΙΕ ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Εκτελεστική Επιτροπή. Τέσσερα λεπτά έχει το λόγο ο κύριος Σάγερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το κοινοβούλιο μας εγκρίνει πάρα πολλές εκθέσεις και εκθέσεις πρωτοβουλίες, οι οποίες εκ των υστέρων φοβάμαι ότι δεν διαβάζονται και από πάρα πολύ κόσμο, αγνοούνται και οι συγγραφείς των προτάσεων αυτών δεν ασχολούνται ούτε αυτοί μαζί τους. Ελπίζω η τύχη της έκθεσης αυτής να είναι διαφορετική. Όχι γιατί την έχω συντάξει εγώ, αλλά γιατί πράγματι συνιστά ένα εγχειρίδιο έλεγα το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους συναδέλφους οι οποίοι σε συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει δημιουργήσει ένα νέο κανόνα ο οποίος αφορά τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα πλαίσια αυτών των νέων κανόνων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει τα ίδια δικαιώματα με το Συμβούλιο σχετικά με τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε βέβαια πάντα τις εκτελεστικές πράξεις όπως επίσης και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Αλλά το κοινοβούλιο μας είναι αυτό το οποίο ε, κατά κάποιο τρόπο ελέγχει τις διαδικασίες αυτές. Όταν σαν παράδειγμα εγκρίνουμε μία νομοθετική έκθεση, στη συνέχεια ε, αγνοούμε την πορεία της εκθέσεως την οποία υιοθετήσαμε στην περίπτωση κατά την οποία δημιουργούνται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά εξουσιοδότηση πράξης. Αυτό ήταν τουλάχιστον αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Από εδώ και πέρα, στα πλαίσια των κατεξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διατηρήσει την επιρροή του, να ασκήσει τα εκτελεστικά τις εκτελεστικές του αρμοδι... να ελέγξει μάλλον τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εκφράσει τη διαφωνία του όταν πράγματι υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε με σωστότερο τρόπο τις αρμοδιότητες τις οποίες εκχωρούμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιες είναι αυτές τις οποίες ασκούμε εμείς σαν κυρίαρχο σώμα. Οι πρακτικές αυτές φυσικά δεν έχουν ακόμα καθιερωθεί πλήρως και οι συνάδελφοι όταν συζητούν στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων με το Συμβούλιο αντιμετωπίζουν μερικές φορές πολλά προβλήματα και διαπιστώνουμε μάλιστα σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το Συμβούλιο εκφράζει μερικές φορές τη δυσαρέσκειά του που έχει χωρίσει κάποιες τέτοιες αρμοδιότητες προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν πράγματι θέλουμε εμείς να υπάρχει σωστός έλεγχος της συνέχεια αυτών των δραστηριοτήτων, θα πρέπει να προβλέπετε μία διαδικασία στα πλαίσια της οποίας δεν μπορεί το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, έλθει, να επανέλθει στα ίδια θέματα εφόσον αυτά έχουν κριθεί από προηγούμενες διαλόγους. Η πρόταση αυτή λοιπόν στην ουσία είναι προσανατολιστική για τους συναδέλφους και τους καλεί να μην παραχωρούν περισσότερα ε, σαρμοδιότητες προς την Επιτροπή. Έτσι θα αποτραπούν καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται, να έχουμε εγκρίνει μία έκθεση με την οποία έχει συμφωνήσει υποτίθεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκ των υστέρων όμως βρισκόμαστε στη θέση να μην μπορούμε να εγκρίνουμε εκθέσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία την οποία προανέφερα. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η επόμενη ε, νομοθετική εντολή να ασχοληθεί με αυτό. Τι είπα. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Σάκια και περνάμε στη διαδικασία Κατσουδιάη. Δίνω το λόγο στην κυρία Μακίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση και αυτά τα τεχνικά ζητήματα, τα συζητάμε σήμερα σε ένα κοινοβούλιο που είναι κενό από συναδέλφους και στην Γεωργία αποσχολήθηκα με το θέμα πάρα πολύ. Δεν έχουμε ακόμη ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση, παρότι εδώ και μήνες ανακοινώνουμε ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά λοιπόν που κάνετε και θα πρέπει αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών που προετοιμάσατε να το διαβάσουν οι συνάδελφοι για να βελτιώσουμε την νομοθετική διαδικασία διαδικασία. Όταν θα καταλήξουμε σε πολιτικές συμφωνίες και πρέπει να περάσουμε τότε στις λεπτομέρειες των πράξεων κατά εξουσιοδότηση των εκτελεστικών πράξεων, θα είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε σωστά. Θα πρέπει από την αρχή να έχουμε διαβάσει το εγχειρίδιο και από την πολιτική γεωργία έχω δει ότι υπάρχουν τρία-τέσσερα δύσκολα ζητήματα που μπορεί μέχρι το Μάρτιο να μην έχουν ολοκληρωθεί, οπότε θα έχουμε πρόβλημα για την υλοποίηση του χρόνου. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η έκθεσή σα από τι πιο σημαντικέ και είναι κρίμα που δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι για να τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ και έχετε δίκιο γιατί είναι μια συνάντηση, μια συζήτηση μεταξύ αυτών που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα μόνο. Η κυρία Βασέσκου. Ευχαριστώ. Οι πράξεις κατεξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις δεν είναι ακόμη σαφές πώς χρησιμοποιούνται. Και γι' αυτό ο ρόλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων θα είναι πολύ σημαντικός και στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Εμείς ως ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε το καθήκον να προστατεύσουμε τους πολίτες της Ευρώπης και να φέρουμε αντίρρηση σε οποιαδήποτε πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αντίθετα προς τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να εμπλέκεται στη διαδικασία πριν από την έγκριση αυτών των πράξεων Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να διοργανώνονται συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν από την έγκριση των πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Ιδιαίτερα σε τομείς όπως η γεωργία, το εμπόριο και τα οικονομικά και νομισματικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Πέρασε τη διαδικασία Σκάτσου και δίνουμε το λόγο στην Επίτροπο Γεωργίευα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Σάιερ για την παρουσίαση στο μικρό αυτό ακροατήριο αλλά και σε αυτούς που μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο τις σκέψεις του που περιλαμβάνονται στην έκθεση αυτή εξ ονόματος της Επιτροπής. Πρέπει να πω σαφώς ότι συμφωνούμε με την ανάγκη να υπάρξει μια κοινή προσέγγιση ό,τι αφορά τις ε, κατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που αναδύονται πολύ συχνά στι διαπραγματεύσει για την ερμηνεία αυτών των κανόνων είναι καιρός να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας για να έχουμε γενικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Η Κομισιόν, όπως ξέρετε, ξεκίνησε τριμερείς συζητήσεις για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή κατανόηση για τα οριζόντια θέματα που άπτονται τον κάθε εξουσιοδότηση και ε, εκτελεστικών πράξεων. Και εκεί τέθηκαν πολλά από τα θέματα τα οποία έχουν αναφερθεί και τονίστηκε η ανάγκη της διαβούλευσης για τις ε, κατεξοδότηση πράξεις Αλλά αυτή η διαδικασία έχει τελματωθεί και χαίρομαι για το γεγονός ότι εσείς δώσατε μια νέα όθηση σε αυτή τη διαδικασία η οποία ελπίζουμε ότι θα μας φέρει σε μια καλύτερη κατανόηση της ε, οριζόντιας αντιμετώπισης των κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με την έκθεσή σα και θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή βάση για να μπορέσουμε να εργαστούμε, για να μπορέσουμε να κλείσουμε την εξέταση των θεμάτων αυτών. Απλώς θα αναφέρω στην προσοχή όλων ότι θα υπάρξει και μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε μια εκρεμή ε, υπόθεση για τα βιοκτώνα όπου το θέμα αυτό των κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων και ελπίζουμε ότι θα μας δώσει και χρήσιμη κατεύθυνση, θα μας δώσει χρήσιμες κατευθύνσεις για τα θέματα αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας για διαδικαστικά θέματα εν ώψη της απόφασης του δικαστηρίου. Αλλά αντίθετα τονίζω ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνεργαστούν για να βρουν <clears throat> αποδεκτές λύσεις για αυτά τα σημαντικά θέματα. Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι σίγουρα το επερχόμενο κοινοβούλιο θα έχει μια πολύ καλή βάση για να επιταχύνει τα, την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων βασιζόμενο στην, στο κοινό έδαφος και στο έργο του κυρίου Σάιερ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Η συζήτηση έχει κλείσει. Η ψηφοφορία θα λάβει και αυτή ε, θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Ευχάριστο βράδυ εύχομαι λοιπόν σε όλους τους συναδέλφους και η φήμη ότι η Κομισιόν δεν κοιμάται ποτέ δεν ευσταθεί απόλυτα.